Colleagues, this colleagues, we have to. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε τώρα, διότι είναι σημαντική η συνεδρίαση και έχουμε πολλούς προσκεκλημένους. Ε, παρακαλώ λοιπόν, καθίστε στις θέσεις σας. Θα περάσουμε στο θέμα 18 στις ε, ατζέντες της Επιτροπής μας. Είναι κοινό θέμα μαζί με τους συναδέλφους ε, της ίντε που είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και χαίρομαι που ήρθε ο συνάδελφος Λάγκη εδώ στο, στο, Προεδρείο, στο Ε, πρόκειται για την επέτειο της τραγωδίας του Ράνα Πλάζα που τώρα ξέρουμε πως λειτουργήσε ως ε, ε, κόδωνας ε, κινδύνου συναγερμού για τον κόσμο της ε, βιομηχανίας ένδυσης. Τόσο για την ΤΕΒΕ όσο και την ΙΝΤΑ έχει πάρει μεγάλη σημασία αυτός ο τομέας γιατί Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα σχέδιο ψηφίσματος πέρυσι που εγκρίθηκε στο, από το Κοινοβούλιο να μας δώσει δεσμευτική νομοθεσία για την δέουσα επιμέλεια και να ζητήσουμε, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για μια δεσμευτική συνθήκη όσον αφορά τα, ε, του ε, τους διεθνείς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρυσι υιοθετήθηκε αυτό το ψήφισμα από την, κυρία, ε, την έκθεση μάλλον της κυρίας Σάντσες και θέλουμε να δούμε τι έχει γίνει έκτοτε από πλευρά της Κομισιόν, αν έχει γίνει οποιαδήποτε, αν έχουμε προχωρήσει προς πιο δεσμευτικό ε, πλαίσιο σε σχέση με την πρωτοβουλία για τον τομέα της ένδυσης. Έχουμε τη Μαριέτα Γιάγκε, προσκεκλημένη ομιλήτρια, που είναι υποδιευθυντής της DG EFCO και είναι συνομιλητής, για μας για το θέμα της βιομηχανίας ένδυσης. Έχουμε τον Μαρίτζιο Λαζάλα που είναι επίσης υποδιευθυντής ε, του γραφείου ε, της ε, του Κέντρου Ανθρωπίνων Πόρων ε, για τις επιχειρήσεις και τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την Μαϊλή Σεσούκε, Γενική Διευθύντρια του οσα του Εθνικού Σημείου Επαφής της Γαλλίας, και εργάζεται για την νέα γαλλική νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας. Έχουμε επίτα τον Βεν Βαν Πέπεστράτ που είναι ε, υπεύθυνο λόμπι ε, και νομικός συντονιστής της εκστρατείας ε, Καθαρά Ρούχα, Clean Clothes Campaign, ΜΚΟ που εργάζεται στον τομέα της ένδυσης όσον αφορά τη βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και δίνω το λόγο στον ε, συνάδελφο Λάγκη. Ευχαριστώ πολύ Λίντα, συμπρόεδρε. Ε, όντως, ε, και οι δύο επιτροπές εξετάζουμε στενά την αξία, την αλυσίδα μάλλον αξίας των αγαθών που έρχονται η πρόεδρος διακόπτη. Παρακαλώ όσοι θέλετε να συνομιλήσετε μεταξύ σας εκτός της αίθουσας. Ε, Ζήτω συγγνώμη, συνάδελφε Λάγκια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποιο που θέλει να ακούσει, μάλλον όσοι ενδιαφέρονται, θα ακούσουν. Εξετάζουμε λοιπόν την αλυσίδα αξία, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι τη σήμερα ημέρα υπάρχουν πολύ λίγα προϊόντα που πραγματικά παράγονται σε μία μόνο χώρα από την αρχή μέχρι το τέλος και γι' αυτό και η εμπορική πολιτική πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην αλυσίδα αξίας και όχι στις ε, συμφωνίες, τις, εμπορ... τις ε, διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε σαφείς ευθύνες, ευθύνες και υποχρεώσεις για τις ίδιες τις εταιρείες ώστε να εντάξουν την διαδικασία της δέσμευσης επιμέλειας στην αλυσίδα παραγωγής. Κάναμε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης, ένα, μια συνεργασία για τα ορυκτά από ζώνες, ε, ε, εμπόλεμες ζώνες ώστε να εξετάσουμε όλη εκείνη την αλυσίδα από το ρηχείο μέχρι την άφηξη αυτών των ορυκτών ε, στην Ευρώπη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και αυτές οι υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι πάνω πάνω στη μέση διάταξη, ειδικά για τον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας πέρα από αυτή την έκθεση που είναι ε, προσανατολισμένη στην αλυσίδα αξιών, εξετάζουμε τις προσωρινές διμερείς εμπορικές συμφωνίες ώστε να κάνουμε μια σαφή δήλωση όσον αφορά το εμπόριο και την βιωσιμότητα, είτε για το κάθε κεφάλαιο, είτε για τις προτιμησιακές εμπορικές ε, ε, συνεργασίες με το GSP, τις γενικευμένες προτιμήσεις και το GSP+. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δούμε τι κάνει η Επιτροπή. Και γι' αυτό και έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας εμπειρογνώμονες. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι οι δηλώσεις τους θα πρέπει να περιοριστούν στα 6 λεπτά εισηγήσεις τους και θα δώσω αμέσως το λόγο στη Μαριέτα Γιάγκερ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι ευρωβουλευτέ, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή ΔΕΒΕ και ΙΝΤΑ. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων περί ενδυση και σα ευχαριστώ που μα φιλοξενήσατε στο, φιλοξενείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πέμπτη επέτειο του τυχήματο τη Ράνα Πλάζα, του που ήταν το πιο θανατηφόρο ε, μέχρι τώρα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα 1.100 θύματα δεν θα ξεχαστούν και ότι τέτοιε τραγωδίες δεν θα να συμβούν στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κυβερνήσει, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους ενδιαφερόμενους φορεί για τις ακούραστε προσπάθειε του προ την επίτευξη αυτού του στόχου. Θέλουμε όλοι να εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια στην αλυσίδα ε, αξία ε, τη ένδυσης και να βελτιώσουμε τη δέουσα επιμέλεια, αλλά και να υπάρξουν πραγματικέ βελτιώσει ε, καθώ και βιωσιμότητα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πω έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος από πολλού φορεί στον τομέα τη ένδυσης τα τελευταία χρόνια. Βεβαίω πολλοί από εμά θα πούμε πω δεν αρκεί η πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά γνωρίζουμε πω. πως οι προκλήσεις ε, του τομέα της Ένωσης όπως τα χαμηλά ημερομίσθια, υπερβολικές ώρες εργασίας, ε, ε, περιορισμένη κοινωνική προστασία, παιδική εργασία, ρήπανση. Υπάρχουν τόσες προκλήσεις όπου πραγματικά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Μας ρωτήσατε τι, κάνει, τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Κομισιόν και φυσικά σεβόμαστε τα ψηφίσματα και τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως οι υπηρεσίες της Κομισιόν καθημερινά συμμετέχουν σε δραστηριότητες με μεγα... πολλούς φορείς ώστε να εξασφαλιστεί πιο βιώσιμη αλυσίδα αξίας. Στον τομέα ανάπτυξης και αναπτυξικής συνεργασίας από που προέρχομαι, αυτό σημαίνει κυβερνήσεις και βασικούς φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να βελτιώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ε, σύμφωνα με τους στόχους της αλλά και σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε πέρσι το Μάιο, δηλαδή χειραφέτηση των γυναικών, αξιοπρεπής απασχόληση, ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια. Άλλη μια απόδειξη για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα στο θεματολόγιο μας είναι ότι θέλω να δηλώσω ότι η ΔΕΦΚΟ αποφάσισε να τοποθετήσει το βιώσιμο ένδυμα στις ε, ημέρες ανάπτυξης που είναι μια εκδήλωση 5 και 6 Ιουνίου σύμφωνα με τις θεματικούς στόχους που είναι φύλλο, ισότητα και χειραφέτηση γυναικών. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι χώροι εργασίας, ε, μάλλον οι περισσότεροι απασχολούμενοι στη βιομηχανία ένδυσης είναι γυναίκες, 75% και επίσης θα γνωρίζετε ε, μάλλον θα είναι εκπρόσωποι και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι ομιλητές αυτή μα την εκδήλωση. Η βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων συμβαδίζει με την, με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Αφρική, ας πούμε, μεγαλώνει η βιομηχανία ένδυσης, ιδιαίτερα στην Αιθιοπία, θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και θα θέλαμε να ε, ε, γίνουν όλα αυτά σύμφωνα με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και είναι αυτό κομμάτι του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου που εφαρμόζουμε, όπου τοποθετούμε την ένδυση, την χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων πολύ ψηλά στο θεματολόγιο. Εάν μου δίνετε, εφόσον μου δίνετε άλλα δύο παραδείγματα ε, λεπτά, θα σας δώσω παραδείγματα για τα προγράμματα συνεργασίας σύμφωνα με τις θεματικές προτεραιότητες. Πρώτη δράση στην οποία βάζουμε πολλά χρήματα, είναι η προώθηση της ε, αλυσίδας αξίας στον τομέα ένδυσης, 65 εκατομμύρια. Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας για την παιδική εργασία και την ε, καταναγκαστική εργασία, βεβαίως ε, ε, και για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασία. Και αυτό είναι σύμμορφο με την ατζέντα μας. Πρόκειται για την έναρξη του προγράμματος το Δεκέμβριο, ανιχνευσιμότητα συνειδητοποίηση και βελτίωση της ε, διαφάνειας. Ε, ένα ακόμα πρόγραμμα που, που στοχεύει την χειραφέτηση είναι η συνεργασία με τον ITC ώστε να ενισχυθεί η, αξία, η αλυσίδα αξίας ε, στην μόδα Μπουρκίνα Φάσο ε, έχουμε ταλαντούχες γυναίκες ε, που προωθούμε στη διεθνή βιομηχανία μόδας. Επίσης προωθείται το περιβάλλον και η βιωσιμότητα από το Switch to Green στην Ασία προς την Αφρική Επίσης εργαζόμαστε σκληρά ώστε να υπάρξει περισσότερη, περισσότερη ενημέρωση για τους καταναλωτές. Έχουμε ένα πρόγραμμα για την ε, συνειδητοποίηση αλλά και για την επανάσταση της μόδας με μια σχετική εβδομάδα εκδηλώσεων και ένα συγκεκριμένο δίκτυ. Επίσης έχουμε και μια ε, υπόθεση ε, ένα πρόγραμμα μάλλον που διευκολύνει τον διάλογο και τις καλύτερες πρακτικές στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των διαφόρων ναυαρχίδων μας ε, όπου η ένδυση είναι μία εξ αυτών. Κάθε εβδομάδα γίνονται συσκέψεις για να μιλήσουμε για την πρόοδο και τις προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει γρήγορη λύση και διόρθωση όλων των προβλημάτων του τομέα της ένδυσης, της βιομηχανίας ένδυσης. Είμαστε προσιλωμένοι στο έργο αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα και να εξασφαλίσουμε πιο δίκαιη και πιο πράσινη βιομηχανία ένδυσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαουρίσιο Λασάλα είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, είμαι από το κέντρο για τις ε, επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλύπτουμε λοιπόν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις σε 180 χώρες στον κόσμο. Την ένδυση την παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό. Πρόσφατα η κυρία Λόλα Σάντζεθ μας ζήτησε μια έκθεση για την δέουσα επιμέλεια των ευρωπαϊκών εταιριών ε, υφαντουργίας. Κυρίως λοιπόν θα σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση που με χαρά μπορούμε να σας τη στείλουμε όταν ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες. Εξετάσαμε 173 απαντήσεις που μας έστειλαν οι επιχειρήσεις από το 2011 από εταιρείε κλωστό υφαντουργίας στην Ένωση για θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αυτό το δείγμα επιστώνουμε ότι 80% από τις κατηγορίες ε, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορούν καταστάσεις σε τρίτες χώρες και σε ποιες περιοχές μάλιστα. Πρώτα απ' όλα στην Ασία 38% των κατηγοριών και κατόπιν είναι οι τρίτες χώρες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία 36% και μετά οι χώρες της Ένωσης 18%. Άλλες περιοχές ε, έχουν πολύ λιγότερες κατηγορίες να τους απευθύνονται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί κυρίως έχουμε ασχοληθεί με την Νότια Ασία μετά το ατύχημα στην Ράνα Πλάζα. Αλλά ακόμη και σε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες, Αλβανία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία και Ουσμπεκιστάν και εκεί η κατάσταση είναι πολύ κακή. Πολύ χαμηλή μισθή, υπερορίες ε, ε, και παρενοχλήσεις των εργαζομένων. Για ποια θέματα θέτουμε ερωτήσεις τώρα. Όπως είπε η κυρία Τζάγκερ, 75% των εργαζομένων παγκόσμια στην ένδυση είναι γυναίκες. Στο Μπαγκλαντές και την Καμπότζη είναι αντίστοιχα 80 και 90%. Άρα δεν μα εκπλήσει που 50% των κατηγοριών αφαιρούν θέματα ισότητα φύλων. Για παράδειγμα, σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Αυτά είναι επιπλέον με τα, με τα γενικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Αυτά είναι τα δύο κυριότερα θέματα που αναφέρθηκαν στο δείγμα μας. Θέματα δηλαδή αμοιβών και επίσης θέματα δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθε. Η ισότητα των φίλων και η ασφάλεια βεβαίω είναι επίση θέματα. Αλλά εμεί κυρίω ασχολούμεθα με θέματα που είναι κάτω από το ραντάρ, που δεν ε, αναφέρονται στα κυριότερα ΜΜΕ. Θέματα που είναι κάπω κρυμμένα και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με μισθούς που να επιτρέπουν να ζήσει, που είναι φυσικά θεμελιώδη δικαίωμα. Το αναγνωρίζει ο διεθνή Οργανισμό εργασία και η Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Και επίση το δικαίωμα να δημιουργία εργατικών ενώσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα, στο Ράνα Πλάζα είχαμε δει ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε συνδικάτο είχαν καλύτερες συνθήκες ε, ασφάλειας και μπόρεσαν να δραπετεύσουν από το κτίριο πιο εύκολα από τους εργαζόμενους που δεν είχαν εκπροσώπηση. Άρα πολλές φορές είναι θέμα ζωής και θανάτου η συνδικαλιστική εκπροσώπηση και η ποιότητα της, ε, των απαντήσεων που μας στέλνουν οι επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, οι περισσότερες εταιρείες δεν μας στέλνουν υψηλού επίπεδου απαντήσεις. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρότερα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρέχουν και αποζημίωση και μέτρα διόρθωσης της κατάστασης. Μόνο 5 από τις 158 επιχειρήσεις που μας απάντησαν με βάση την ε, γνωστή μεθοδολογία για την παρουσίαση θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μόνο λοιπόν πολύ λίγε επιχειρήσει μα έστειλαν υψηλού επίπεδου απαντήσει. Πολλά πρέπει να γίνουν. Επίση, υπάρχουν θέματα σύγχρονη δουλεία και πώ την αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει. Υπάρχει για παράδειγμα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο Πρέπει λοιπόν και στο G7 και στο G20 να αποκτήσουν περισσότερη προτεραιότητα τα θέματα αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των διαφόρων ε, επιχειρήσεων του κλάδου. Για παράδειγμα, το Adidas ε, έχει 81% στην κλίμακα για την ε, σύγχρονη δουλεία ενώ η εταιρεία Brother ε, είναι μόνο στο 9%. Ευρύτατο το χάσμα δηλαδή μεταξύ διαφόρων εταιριών στην κλωστοεφαντουργία στην Ευρώπη. Εξετάζουμε τώρα και τις δικαστικές ε, αποφάσεις και δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά, αλλά όλα μας τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και δεσμευτικής νομοθεσίας, ούτως ώστε να υπάρξει δυνατότητα ενδίκων μέσων για τα θύματα για να ε, προωθηθούν οι ηγέτες και να ευνοηθούν και να καταλάβουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν εύκολα τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργείται συνθήκες για μια προσπάθεια εναρμόνισης προς τα πάνω. Πρέπει να αναρμονιστούν οι πρακτικές και να αποφύγουμε διάφορες ερμηνείες, ε, τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων για μη οικονομικά θέματα και τις γερμανικές και ολλανδικές πρωτοβουλίες που σύναψαν ένα σύμφωνο. Και ε, οι εθελούσιες ε, πρωτοβουλίες έχουν περιορισμένο αποτέλεσμα. Δεν αντιμετωπίζουν τα συστημικά θέματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε όμως τι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ για τα κλώστο υφαντουργικά. Θα μπορούσε να είναι η βάση για δεσμευτικές υποχρεώσεις προ τι επιχειρήσει. Και στη Γαλλία υπάρχει και αυτός ο νέος νόμος για την δέουσα επιμέλεια από τις μεγάλες εταιρείες. Και τώρα από το σημείο επαφής για τη Γαλλία η κυρία Μαλέ Τσάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θυμίσω γαλλικά, παρακαλώ να έχουμε και το και της διαφάνειες Είμαι Μαϊλή Σουκ, Γενική Γραμματέας του Εθνικού Σημείου Επαφής της Γαλλίας για την υπευθυνότητα των εταιριών που θέλει ακριβώς να εφαρμόσει αυτές τις αρχές στη Γαλλία. Σε 5,5 λεπτά είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσω αυτά που κάναμε μετά το δράμα του Ράνα Πλάζα. Τρεις εβδομάδες μετά το δράμα αυτό, η Γαλλίδα Υπουργό του Εξωτερικού Εμπορίου απευθύνθηκε στον οργανισμό μας για να εξηγήσουμε τι συνέβη με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Και στο Δεκέμβριο του 2013 υποβάλαμε στην Υπουργό μια έκθεση που εξηγεί πολύ συγκεκριμένα τι σημαίνει λογική δέους επιμέλεια και ευθύνη των πολυεθνικών στις αλυσίδες προμηθειών της παγκόσμιας κλώστου εφαντουργίας. Πολύ σημαντική έκθεση. Η Υπουργός υιοθέτησε όλες μας τις συστάσεις και κατόπιν ζήτησε από τον οργανισμό μας να παρακολουθήσει την κατάσταση και να στείλει τα αποτελέσματα στον ΟΣΑ. Εμείς στην έκθεσή μας πρώτα απ' όλα εξηγούσαμε τις αλυσίδες προμήθειας, τις παγκόσμιες και καταλήξαμε σε πορίσματα πολύ παρόμοια με τους προηγούμενους, παρουσίαζε τις αλυσίδες και έκανε διάφορες συστάσεις και στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές λόγω της περιπλοκότητας ε, των προβλημάτων και της ανάγκης συλλογικής, συντονισμένης, πολυμερούς και διεθνούς αντιμετώπισης. Και τι έχει συνέβη έκτοτε. Το γαλλικό PSN, όπως λέγεται ο οργανισμός μας, παρακολουθεί την εφαρμογή της έκθεσης στη Γαλλία, παρακολουθήσαμε τη συμφωνία με το Μπαγκλαντές, τις ε, πρωτοβουλίες των Διεθνών ΜΚΟ και των Διεθνών Οργανισμών Συνδικάτων. Συναντηθήκαμε με διάφορους επικεφαλείς και φτιάξαμε μια γαλλική ομάδα για την υπεύθυνη αλυσίδα προμηθειών που είναι η γαλλική εκδοχή των ε, γερμανικών και ολλανδικών πρωτοβουλειών που μόλις αναφέρθηκα. Εγώ ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τη λειτουργία αυτής της γαλλικής ομάδας εργασίας που στόχο έχει να υπάρχει ευρύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων του PSN από τις γαλλικές επιχειρήσεις και επίσης καλούμε εκπροσώπους του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ ή και του CCC, ούτω ώστε να καταλάβουν και οι Γάλλοι τις εξελίξεις και πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, στα πλαίσια του ΟΣΑ αναπτύξαμε δράση. Από το 2014 υπάρχει μία ομάδα που ασχολείται με τις αλυσίδες παραγωγής και την εφαντουργία, και μετά από επίπονη πολιτή εργασία πέρυσι το 2017 ο ΩΣΑ υιοθέτησε αυτό τον οδηγό για την υπεύθυνη αλυσίδα προμηθειών που ενισχύει την έκθεση του ΠΣΕΝ είναι θεμελιώδης εργασία πολυμερής, διεθνής σημείο αναφοράς πολύ σημαντικό επιπλέον, επιπλέον συγγνωμιώσα δημιούργησε αυτόν τον οδηγό υπάρχει το Παγκόσμιο Φόρουμ για την κλωστοεφαντουργία που συνεδριάζει κάθε χρόνο και φέτος θα ασχοληθεί με δύο πολύ σημαντικά σημεία που συζητήθηκαν. Το πρώτο είναι πολύ τεχνικό. Είναι μια, ένα εργαλείο για τον συντονισμό των πρωτοβουλίων γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Μέσω αυτού του εργαλείου που είναι στη διάθεση όλων μπορούν να ελέγξουν εάν υπάρχει λογική επιμέλεια. Είναι εντελώς νέο μπήκε στο site του ΟΣΑ πρόσφατα και επίσης υπεγράφει μια εταιρική σχέση μεταξύ του ΟΣΑ και του ΣΕΝΤΑΚ που είναι η μεγαλύτερη κινέζικη εξαγωγική εταιρεία προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους ε, Κινέζους εταίρους μας για να υπάρχουν ε, οι αναγκαίες τυποποιήσεις συμμετέχει ο οργανισμός αυτός από 14 εργασίες μας. Κάτι άλλο. Μας στηρίζει συνεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σημαντικό. Χρηματοδοτεί τις εργασίες του ΟΣΑ. Αλλά όπως μόλις είπε η κυρία αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, αναπτύσσει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τον ΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας για να εφαρμόζονται οι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργαζομένων επιτόπου. Ορίστε λοιπόν πώς ε, λειτουργεί ο ΩΣΑ. Και πέρα από όλα αυτά, στη Γαλλία, κάναμε πάρα πολλά για το νομοθετικό πλαίσιο. Ξέρετε, εγκρίναμε ένα νέο νόμο κατά της διαφθοράς το 16 και το 17 ε, το νόμο για την υποχρέωση επαγρύπνησης και επίσης ε, ένα νέο διάταγμα για την υποβολή μη οικονομικών εκθέσεων και καταλαβαίνουμε ότι όλη η εργασία που έχει κάνει το PSN για την γλωσσική φαντουργία και όλη η εργασία που έγινε στον ΩΣΑ θα μας βοηθήσουν στην εφαρμογή αυτού του νόμου. Καταλήγω λοιπόν στη συμπληρωματικότητα των μέσων ε, αυστηρού και υπείου δικαίου για όλους τους συμμετέχοντες και Μόνο πολυμερός, μόνο συλλογικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στην κλωστοφαντουργία. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Βέβαια, πολλά συνδικάτα και εμεί κυβερνητικές οργανώσεις ασκούν πιέσεις για ακόμα περισσότερες βελτιώσεις στην κλωστοφαντουργική βιομηχανία και οι εκπρόσωποι μιας από τις πιο σημαντικές ε, ε, οργανώσεις είναι ο κύριος Βαντεστράτε, ο οποίος είναι παρόν εδώ και του δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, για να σας ε, απευθύνουμε το λόγο. Πάντοτε με ευχαρίστηση έρχομαι εδώ στον οίκο τη Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να συμβάλλω και εγώ στην συζήτηση του θέματος αυτού και ιδίω τώρα, σήμερα, μια πενταετία μετά από το συμβάν στη Ράνα Πλάζα, που είναι μια σωστή ευκαιρία για να σκεφτούμε ποια πράγματα έγιναν μετά και ποια δεν έγιναν. Σύντομα λίγα επιτεύγματα που ε, έχει να, δείξει, να επιδείξει ο τομέας συνολικά. Πρώτο και πιο σημαντικό, ότι μπορέσαμε να ε, προσφέρουμε ρύθμιση για επανορθώσεις στα θύματα ε, οικονομικές αποζημιώσεις δηλαδή στα θύματα της Ράνα Πλάζα, κάτι το οποίο έκαναν πραγματικότητα όλα τα μέρη μαζί. Το ατυχές εδώ είναι ότι εν τέλει με τη συλλογή κονδυλίων χρειαζόταν και κάποια πίεση εκ των άνω για να δοθεί η οικονομική επανόρθωση στα θύματα. Χρειάζεται λοιπόν να μπουν οι ράγες ώστε να είναι πιο μόνιμο το σύστημα Το δεύτερο που επιτύχαμε ήταν η συμφωνία για την πυρασφάλεια στο Μπαγκλαντές, αυτό αναφέρθηκε ήδη, πρόκειται για ένα σύμφωνο μεταξύ παγκόσμιων φορέων και τοπικών φορέων, ε, μη κρατικών οργανώσεων και αρμόδιων αρχών, που δεσμεύονται να επιθεωρούν τα εργοστάσια για ζητήματα πυρασφάλειας και όταν εντοπιστούν σχετικές ελλείψεις να τις διορθώνουν και αναλαμβάνουν και τη δέσμευση να ε, δώσουν και τα σχετικά κονδύλια εφόσον υπάρχει ε, θέμα χρηματοδότησης. Πέντε χρόνια μετά λοιπόν 85% περίπου των θεμάτων έχουν επιληθεί, παραμένουν όμως κάποια ζητήματα ανοιχτά και γι' αυτό ως ε, οργάνωση που διεξάγουμε εκστρατείες προχωρούμε δεύτερο σύμφωνο με 145 συμβαλόμενα μέρη όπου να περιληφθούν και άλλες ε, βιομηχανίες, ε, να ε, ασχοληθούμε και με θέματα ελευθερίας του συνεταιρίζεστε και βέβαια και με την σεξουαλική ή γενετήσια παρενόχληση, η οποία είναι ένα σημαντικό θέμα στα εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας του Μπαγκλαντές. Η συμφωνία πάντως εργοστασια κλωστοφαντουργιας μαρτυρία ότι μία προσέγγιση με ξεκάθαρες δεσμεύσεις και κανόνες και λογοδοσία για τους κανόνες αυτούς αποδίδει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν κάποιο νόημα για τους εργάτες και τις εργάτες επιτόπου. Πρώτο που μας απασχόλησε ήταν η αυξημένη διαφάνεια, διότι υπάρχει μεγάλη διαφάνεια στον ε, κλάδο. Έχουμε δημοσιεύσει τις, τα αποτελέσματα των εκθέσεων, λίστες ε, ε, των συμμετεχόντων και των ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί. Με την έννοια αυτή η διαφάνεια ε, βοηθά και την συμμόρφωση. Η διαφάνεια είναι το τρίτο επίτευγμα του κλάδου, διότι σύμφωνα και με τα όσα προβλέπει η συμφωνία, εμείς μαζί με άλλους φορείς ε, της κοινωνίας των πολιτών όπως η Human Rights Watch και άλλοι οργανισμοί πιέζουμε τον κλάδο ε, να δημοσιεύει ε, τα ονόματα εργοστασίων που δεν έχουν συμμορφωθεί και μάλιστα ορισμένα που θα έχουν κλείσει. Ταυτόχρονα παραμένουν πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει ακόμα να διορθωθούν. Στο Μπάγκλατες και μόνο οι μισθοί παραμένουν πρόβλημα. Η αγοραστική δύναμη των μισθών είναι μάλιστα χαμηλότερη από ό,τι προ πενταετίας. Η ελευθερία του συνεταιρίζεστε παραμένει θέμα. Τα συνδικάτα εξακολουθούν να διώκονται ε, σε πολλά μέρη του κόσμου και στο Μπαγκλαντές ακόμη. Όπως είπα, η γενετήσια παρενόχληση παραμένει ε, παρούσα σε μεγάλο μέρος του κλάδου. Αυτά για την Μπαγκλαντές, όπου έχουμε και ειδικό μηχανισμό για τη λογοδοσία EPA Trade Preferences. Είναι γενικότερο όμως το κακό αυτό στην κλωστοεφαντουργία. Η συνάδελφός μου μίλησε προηγουμένως για χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάτες και εργάτριες της κλωστοϊφαντουργίας που λαμβάνουν μισθούς παρόμοιους με αυτές των Παγκλατεσιανών. Όταν λέω ότι πολλά ακόμα μένουν να γίνουν, μιλώ για τέτοια πράγματα. Πρόκειται για πραγματικά μεγάλο έργο για να ε, επέλθουν βελτιώσεις στη ζωή των εργαζόμενων επιτόπου. Έτσι, με την έννοια αυτή, νομίζω ότι αφενός δείχνοντας ότι ένα καθεστώς λογοδοσίας αποδίδει από την άλλη μεριά ότι μένουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα από την κλωστοϊφαντουργία, σας ενθαρρύνουμε εσάς ως ευρωβουλευτές να στοχεύσετε σε κάποια θέματα που θα μπορούσαν για τα επόμενα χρόνια να είναι να προωθήσετε αυτά που ζητεί το ψήφισμα για την δέουσα επιμέλεια των ε, κλωστοϊφαντουργικών βιομηχανιών, να βασιστείτε στο έργο του ΟΟΣΑ, που το υποστηρίζετε και αποτελεί σωστή βάση και να υποχρεώσετε τις επιχειρήσεις να εξετάζουν τι γίνεται μέσα στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και όταν εντοπίζονται θέματα να αρχίσει και μια προσπάθεια διόρθωσής τους και να αναλαμβάνονται οι ευθύνες για ενδεχόμενες επιπτώσεις. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, ακούσαμε τέσσερις εμπειρογνώμονες. Ίσως ε, αναφύεται η ερώτηση γιατί δεν είναι παρούσα η ίδια η βιομηχανία. Ε, ο εκπρόσωπος ε, το, της αλυσίδας CNTA δεν είναι ακόμη εδώ λόγω... Αλλά έρχεται τώρα, λέει η κυρία Μακάβαν. Τώρα μόλις μπαίνει στο κτίριο. Μόλις έρθει θα του δώσουμε το λόγο όταν θα φτάσει εδώ. Είναι ζήτημα καθυστέρηση του ταξιδιού του. Έτσι ώστε να υπάρχει κάποια σοβαρή εκπροσώπηση. Να δώσω τώρα το λόγο πάλι στην Ελίντα Μακάβαν που είναι η συμπροεδρός μου Μάλιστα, ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και ξεκάθαρα μηνύματα για το τι μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτέ σχετικά. Να ακούσω πρώτα την Λόλα Σάντσε, που είναι η εισηγήτρια για την εμβληματική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, κλάδο τη κλωστοϊφαντουργία. Λόλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ε, Λίνα, και ευχαριστώ πολύ και τους ομιλητές που ήταν σήμερα εδώ θα ήταν καλύτερα να έχει έρθει στην ώρα του ο εκπρόσωπος ε, της βιομηχανία, γιατί όταν έρχεται η στιγμή, χθε ας πούμε στο Twitter, εγώ, τοποθε... εγώ έβαλα κάποια post στο Twitter και στη συνέχεια Βγήκε η Ζάρα, η εταιρεία Ζάρα να μου απαντήσει ότι δεν είχε σχέση με τη Ραναπλάσα και ότι δεν ήταν καν εκεί. Εγώ συνεχίζω τη συζήτηση γιατί αυτό που θέλω είναι να έρθουν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο να καθίσουμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε μια πιθανή μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ωφελούσε όλου. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω είναι να κάνω αυτή την δημόσια έκκληση προ την εταιρεία Inditex να έρθει εδώ. Δεν, ε, με το που το είπα αυτό δεν μου απάντησαν πια. Τελείωσε η συζήτηση. Το ναι, ούτε όχι. Όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας, αυτές οι μεγάλες εταιρείε τι κάνουν, εξαφανίζονται. Δεν δείχνουν το πρόσωπό τους. Εγώ δεν είμαι εχθρός, ούτε θέλω να είμαι εχθρό. Θέλω να καθίσουμε, να συζητήσουμε μαζί και να βρούμε κοινά σημεία που θα εφελήσουν όλους. Θα είμαι σύντομη, αλλά θα ήθελα να θυμίσω κάτι που κάποιες φορές ε, ε το ξεχνάμε. Είναι η καταστροφή αυτή ή το έγκλημα που έγινε, συνέβη στη Γαλλία, στην Κουριέρ, κοντά στην, στα σύνορα με το Βέλγιο, το 1906. Ε, ε, πήρε φωτιά ε, όπου δούλευαν πάνω από 1500 άνθρωποι τότε εκεί και παιδιά και η εταιρεία προσπάθησε να σώσει ε, διάφορους, αλλά ε, η προτεραιότητα ήταν παρόλα αυτά να διατηρηθεί το ορυχείο και να σωθεί το, το ορυχείο. Και τι κάνανε, φράξαν τις εξόδους ε, του ορυχείου για να α, α, σβήσει φωτιά. 1099 έχασαν τη ζωή τους εκεί μέσα. Αυτό έγινε το 1906. Μας φαίνεται κάτι πολύ μακρινό. Όμως αυτό που έγινε στο Ρώνα Πλάζα είναι πολύ παρόμοιο. Το 1906 όμως ξεκίνησε η ενώση ε, των ε, ε, ανθρακορίχων και τότε στη Γαλλία φτιάχτηκε το πρώτο Υπουργείο Εργασίας του κόσμου και ο πρώτος κώδικας εργασίας στον κόσμο. Ήταν η πρώτη νομοθεσία που αφορούσε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ουδέν κακό να μηγές καλού όπως λέμε. Μετά από την καταστροφή στο Ράνα Πλάσα, πέντε χρόνια αργότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιστάσεις για να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να τι να κάνουμε για να συζητήσουμε πώς θα τοποθετήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Πράγματα τα οποία ζητάμε δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια. Η παγκοσμιοποίηση δεν, ε, δεν με βρίσκει σύμφωνη, αλλά συμβαίνει. Είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε κριτήρια, ε, να μπορούν οι εταιρείε μας να μπορούν να λειτουργούν, αλλά κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια με τους δικούς μας συμπολίτες, θα πρέπει να επιτρέπουμε να γίνεται ούτε και αλλού, γιατί διαφορετικά είναι πολύ κοινική αυτή η ε, στάση. Αυτό βλάπτει την εικόνα μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δείχνει και την, ε, δίνει λαβή στο να επιτεθεί κανείς ε, στις ευρωπαϊκές αξίες που ωστόσο οι πολίτες εξακολουθούν να υπερασπίζονται. Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργεί ο κόσμος ε, της μόδας. Όλοι θα συμφωνούσαν να πληρώσουν λίγο παραπάνω ή ε, εν πάση περιπτώσει να υπάρχει καλύτερη σήμανση στα ρούχα ώστε να μπορεί κανείς να διαλέξει γνωρίζοντας τι συμβαίνει. Τώρα, υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Πάρα πολλέ εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνουν ε, τα τελευταία δέκα χρόνια. Άγριο ανταγωνισμό. Πώ τον καταμολυμούν, ε, επενδύοντα στην ποιότητα υψηλού επίπεδου επενδύσει. Και υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα, ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος της πιστοποίησης, ότι όντως κάνουν τα πράγματα σωστά. Οπότε τελικά το κόστος αυτό έχει αντίκτυπο. Στο ποιο το κάνει καλύτερα, ποιος αυτός που το κάνει χειρότερα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται να δώσει καμία εξήγηση. Τα όσα όμως γίνονται εδώ, αυτοί που λειτουργούν εδώ και θέλουν να λειτουργήσουν ποιοτικά και να έχουν το πιστοποιητικό ποιότητας, ε, πληρώνουν μεγαλύτερο κόστος γιατί έτσι το απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, απλώς να επιμείνω. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από το ατύχημα του Ραναπλάσα, αλλά καθημερινά υπάρχουν προσωπικά ατομικά ε, χιλιάδων ανθρώπων που υποφέρουν ε, στη ζωή τους για να μπορούν εμάς να μας δίνουν. Ε, αυτά και ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, ευχαριστώ που ήρθατε. Υπάρχει το άνοιγμα, πρέπει απλά να, να μπορέσουμε να πιέσουμε ώστε όλα αυτά τα λόγια να γίνουν και πράξεις. Ευχαριστώ. Θέλετε να πάρετε αμέσω το λόγο, απευθύνεται η πρόεδρο στον ομιλητή από το CK. Στον ομιλητή από το CK. Ναι, αφήστε με να πάρω μια ανάσα παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, βουλευτέ. Η πρώτη ομιλητρία είναι η Άγνες Γιονγκέριους. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Γιατί ίσως θα μπορούσατε κι εσείς να μιλήσετε για αυτό το ε, θέμα που με απασχολεί. Πέντε χρόνια μετά από το Ράνα Πλάζα και ένα χρόνο μετά την έκθεση, εδώ στο, την κατάθεση αυτής της έκθεσης μάλλον εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, βλέπουμε κάποια πρόοδο. Και είμαι ικανοποιημένη από τα θετικά παραδείγματα που αναφέρατε, αλλά έχω μια απορία. Πρώτον, η με τα οποία να μπορεί κανείς να ζήσει. Και βλέπω και τον εκπρόσωπο του CK. Τι θα γίνει με τα κέρδη σας ή τα περιθώρια κέρδους σας αν ο κόσμος στο Μπαγκλαντές ή και αλλού ε, ο κόσμος που εργάζεται δηλαδή στον τομέα της ένδυσης μπορούσε να κερδίσει ένα, ε, αξιοπρεπή μισθό με τον οποίο μπορεί να επιβιώσει. είναι πιθανό πέρα από τις ρυθμίσεις για την σεξουαλική παρενόχληση ε, να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείε ώστε να υπάρξει πίεση για, μια, για έναν ε, μισθό διαβίωσης και η επόμενη με ερώτηση απευθύνεται στην DG DEFCO. Ειδικά για την περίπτωση του Μπαγκλαντές, εσείς μαζί με συναδέλφους του DG Ample και Trade είχατε στείλει δύο προθεσμίες στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές προσπαθώντας να τους αναγκάσετε να ξεκαθαρίσουν τα νομοσχέδια περί εργασιακής νομοθεσίας. Έχουμε όμως πάλι μια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου εργασία για τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης. Πότε λοιπόν θα προβείτε στα επόμενα βήματα προς την ε, κυβέρνηση, ε, τι διαβήματα θα κάνετε προς την κυβέρνηση του Παγκλαντές, γιατί αν θέλουμε να παίρνουμε τον αυτό μας σοβαρά, ε, υπόψη. Εφόσον υπάρχουν δύο προθεσμίες, τις αφήνουμε να περάσουν και δεν κάνουμε τίποτα, χάνουμε την αξιοπιστία μας. Τι προτίθεστε να κάνετε λοιπόν, τι διαβήματα προ την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ. Ε, μάλιστα, πολλοί ακόμα ζητούν τον λόγο. Έχουμε ακόμα δύο ομιλητέ. Παρακαλώ, μάξιμουμ δύο λεπτά έκαστος. Ίσως καλύτερα να πάρετε τον λόγο μια και καλή στο τέλο να ακούσετε τι ερωτήσει, ώστε να μπορέσετε να προσθέσετε κάτι στην ομιλία σας. Μάξιμουμ δύο λεπτά θα είμαι πολύ αυστηρή γιατί ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί σε διάφορα επίπεδα, ιδιαίτερα από πλευρά ΜΚΟ και ΩΣΑ. Μόνο μερικά παραδείγματα που ήδη τα παρουσίασαν πολύ καλά οι ομιλητέ μα. Αλλά αυτέ οι πρωτοβουλίε είναι μια αντίδραση στην έλλειψη αντίδραση των αρχών και της πολιτικής για να καλυφθούν τα κενά, οι αποτυχίες της διεθνούς κοινότητας να αδράξει το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν καθαρά πολιτικό θέμα και θέμα διακυβέρνησης. Όταν βλέπουμε ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη διακυβέρνηση, έχουμε την ΚΝΟΥΣΕΝΤ, το Διεθνή Οργανισμό εργασία, το Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, τον ΟΣΑ. Αυτοί συνεδριάζουν τακτικά είτε σε επίπεδο πρέσβεων, είτε σε επίπεδο υπουργών. Υπάρχουν και εκπρόσωποι υπουργείων σε όλε αυτέ τι συνεδριάσει. Αλλά Νομίζω ότι είναι σαφές ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο συμμετοχής σε αυτές τις συζητήσεις, ε, τόσο καλύτερες είναι οι αποφάσεις. Για παράδειγμα, γιατί να μην πάει στο G20, όπου συμμετέχουν και οι βιομηχανικές χώρες και οι αναπτυσσόμενες και υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς, ως ε, πολιτική ομάδα, θα πρέπει να φροντίσουμε να εγγραφεί στην ημερή διάταξη του G20 το θέμα αυτό. Είχα γράψει μια επιστολή στην κυρία Μέρκελ πριν από ένα χρόνο όταν προέδρευε στο G20 καλώντας την να το θέσει στην ημερήσια διάταξη. Το ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές προδιαγραφές στον κλάδο. Και μου απάντησε ότι είχα καθυστερήσει. Δεν υπήρχε πλέον χρόνος. Δεν προλαβαίνανε πια για, για πέρυσι. Ε, ας το βάλουν φέτος σε όλες τις ημερήσεις διατάξεις του G20 στο μέλλον θα πρέπει να μπαίνει. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε να αλλάξουν τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο. Όλες οι πρωτοβουλίες που αναφέρθηκαν είναι θαυμάσιες, κρίσιμες, απαραίτητες, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να ε, απέχει η πολιτική. Η Άννη Λίτς. Ο, ο κύριος Λίτς Ευχαριστώ τις δύο επιτροπές χθες ως πρόεδρος στο Χάλε ήμουν παρόν σε μια επανάσταση της μόδας όπου συμμετείχε και ο ΩΣΑ και πρέπει να εξετάσουμε και την υπόδειση, όχι μόνο την ένδυση και τα δερμάτινα όλα αυτά ανήκουν στον ίδιο κλάδο δεν έχουμε εισακουστεί από την Κομισιόν. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον κύριο Τίμερμαντ. Ο κύριο Νίμιτσα είχε πιο ανοιχτή προσέγγιση. Αλλά ποτέ δεν του συναντήσαμε και του δύο μαζί. Δεν με ικανοποιεί αυτό. Ενδιαφέρεται η Κομισιόν να ασχοληθεί. Δεν παίρνει σοβαρά το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δεν θα υπάρξει νομοθετική προσέγγιση. Δεν θα μπορούσαμε φέτος να ξεκινήσουμε μια πλατφόρμα που να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με βάση την γερμανική και ολλανδική πρωτοβουλία, ώστε να συμμετέχουν όλοι. Έτσι θα προχωρήσουμε με βάση τι προδιαγραφέ στην Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία. Επίσης, υπάρχουν νέε εξελίξεις στο Μπαγκλαντές. Όταν ε, είχαμε πάει εκεί, με βάση την πρωτοβουλία όλα εκτός από τα όπλα κάναμε ορισμένε προτάσει. Ποια είναι η αντίδρασή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Μαρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά τραγικό ότι πρέπει πρώτα να συμβεί μια καταστροφή για να αρχίσουμε να αντιδρούμε. Και το 1906 μας θύμισε η Λόλα πώς ήταν τότε και τα πράγματα πάλι παρόμοια είναι σήμερα. Εμείς βλέπουμε τις άσχημες αυτές καταστάσεις εδώ και πολλά χρόνια και κοινωνικά και οικολογικά. Στην έκθεσή σας, ή τέλος πάντων στην αρχική σας παρέμβαση, είπατε ότι υπάρχουν ακόμη ελλείψεις και στα οικειοθελή μέτρα. Εμείς μιλούμε όμως εδώ και κυρίως για τις ελλείψεις της νομοθεσίας. Ερώτηση λοιπόν, όπως λέτε στην έκθεσή σας, εξετάσατε πώς λειτουργούν τα οικειοθελή μέτρα. Η Γερμανία έχει κάνει κάποιες ρυθμίσεις ε, δημιουργώντας αυτό το δίκτυο της ε, δίκαιης ευκλωσιβαντουργίας. Όλα αυτά έμειναν όμως μέσα στον τομέα των οικειοθελών μέτρων. Καλά είναι αυτά, αλλά χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Έχετε αξιολόγηση κατά πόσον ε, απέδωσαν αυτά τα οικειοθελή μέτρα ή προχωρούν κάποια βήματα και μετά βέβαια τους φαίνεται το κέρδος σημαντικότερο από τις ζωές των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Και όπως είπε ο Σαρλ Γκέρενς προηγουμένως, στην πολιτική έχουμε σημειώσει σημαντικές παραλήψεις τις οποίες πρέπει να καλύψουμε γιατί δεν μπορεί η βιομηχανία να αυτοπεριορίζεται ή να αυτορυθμίζεται και ο θελός και κάποια στιγμή να σταματά. Ο νομοθέτης πρέπει να δράσει. Νόιζερ. Ευχαριστώ. Έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων μου από τις προηγούμενες ε, συναδέλφους μου. Θέλω να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έγινε τον τελευταίο χρόνο. Είχαμε πάει το Μάρτι πέρσι εκεί. Είχαμε ακούσει πολλά για προθεσμίες στο Μπαγκλαντές. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν, ποιε βελτιώσει επιτεύχθηκαν τελευταία, τον τελευταίο χρόνο μάλλον, ε, ειδικώ για τον Μπαγκλαντές. Πρόεδρο. ωραία. Α, ακόμα μία συνάδελφος, μάλιστα. Η κυρία Μινέρ. Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Ολλανδικά όχι, ε. Μπορώ να μιλήσω και Ολλανδικά. Βεβαίω, να, τόσοι διερμηνεί εδώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, λοιπόν, το δράμα αυτό της Ρανά Πλάζα μετά από αυτό το δράμα η Κομισιόν ε, ανέλαβε πρωτοβουλίες και με τις τοπικές αρχές αλλά και με τον ε, Διεθνή Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας. Η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες και ε, για παράδειγμα σε άλλες χώρες όπως το Σριλάνκα ή το Πακιστάν. Αυτά τα UN Guiding Principles τα οποία περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά ε, απευθύνονται και σε επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τι γίνεται τώρα με την υποχρέωση ιδέουσας επιμέλειας. Εάν δηλαδή είναι προφανές ότι χάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι άνθρωποι μπορούν να προσφύγουν. Υπάρχει τρόπος να προσφύγουν ε, δικαστικά. Γιατί συχνά υπάρχουν... Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Λίντα Μακάβαν, ο κύριος Κονσάλες από το C&A, επειδή ε, με κάποια καθυστέρηση δεν πρόλαβε να μιλήσει. Ίσως θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για την παρουσίαση που είχατε ετοιμάσει, αλλά και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Λυπούμε που καθυστέρησα, δεν οφείλεται στην ισπανική μου κουλτούρα. Ε, υπήρχε ε, κάποια διαφορά μεταξύ της γραμματείας μου και μου σε ό,τι αφορά ε, τις ε, υποχρώσεις μου. Ε, δεν είχα καν παρουσίαση. Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να παρουσιάσω, ούτε καν ολόκληρο βέβαια, τον κλάδο. Ο κλάδος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ευρύτατος. Υπάρχουν πολλές μάρκες, πολλές οργανώσεις που παράγουν κλωστεφαλαιτουργικά προϊόντα απανταχού του κόσμου. Η C&A δεν εκπροσωπεί βέβαια όλον τον κλάδο. Η εκπροσωπεί τι οργανώσει οι οποίε πιστεύουν σε πραγματικέ αληθινές αξίε και ενδιαφέρονται να αλλάξουν τα πράγματα στην ε, αλυσίδα προμήθεια ή προμηθειών. Και όταν μιλούμε για τον αριθμό αυτό ε, ε, εταιριών ή οργανώσεων ή μάρκας, είναι μια χούφτα αυτές που τα κάνουν αυτά και αποτελεί πρόκληση και για μας όταν εμείς ως μάρκα ερχόμαστε να συζητήσουμε με εργοστάσιο ή με προμηθευτή όπου εκεί παράγουν και άλλες μάρκες, αυτό είναι πρόκληση και για μας, για να διατηρήσουμε τις αξίες μας σε υψηλό επίπεδο. Εδώ εκπροσωπώ, θα έλεγα, τις οργανώσεις εκείνες οι οποίες έχουν ε, υπογράψει, για παράδειγμα, το Σύμφωνο του Παγκλαντές. ή εκπροσωπώ τις οργανώσεις εκείνες οι οποίες έχουν συνυπογράψει το μνημόνιο ε, κατανόησης για ε, τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Υπάρχουν πολλοί, πολλές οργανώσεις, πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν κάνουν τέτοια πράγματα όπως το CNT για να αλλάξουν την ε, βάση προμήθειας. Και έτσι όμως θεωρούμε και εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Προπενταετίας έγινε αυτό το τραγικό ατύχημα στο Ραναπλάζα. Η C&A έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια από την αρχή να βρει τι καλύτερε δυνατές λύσεις και άλλες βεβαίω οργανώσεις ή άλλες επιχειρήσεις. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη το ατύχημα αυτό ήταν διότι υπήρχαν κακές πρακτικές σε διάφορους τομείς και από την ε, ε, πλευρά της επιχειρήσης και από την πλευρά της κυβέρνηση του Μαγκλαντές και ε, κακέ πρακτικέ, ασφαλμένε πρακτικέ και από άτομα επιτόπου. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά είναι με συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν κάποιες αλλαγές. Και με τα UN Guiding Principles που είμαι βέβαιο ότι τα γνωρίζετε όλα, αυτά τα Guiding Principles ξεκαθαρίζουν ποια είναι τα στοιχεία που είναι ευθύνης των επιχειρήσεων. Αλλά καθορίζουν και πού αλλού εντοπίζονται οι ευθύνε κυβερνήσει. Και όταν μιλώ για κυβερνήσεις, μιλώ για όλους τους κυβερνητικού φορείς οι οποίοι μπορούν να θεσπίζουν νομοθεσία αλλά και να φροντίζουν για την εφαρμογή της. Δηλαδή περιλαμβάνω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για το λόγο αυτό βρίσκομαι άλλωστε εδώ, διότι και εσείς φέρετε ευθύνη και βεβαίω θέλετε να ε, ε, αναλάβετε τι ευθύνε αυτές. Ε, υπό την έννοια αυτή Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία τα οποία στηρίζουν την αύξηση ή βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, των συνθήκων εργασίας στην, στην ε, αλυσίδα προμηθευτών. Εμείς έχουμε περιορισμένη ικανότητα να επιφέρουμε αλλαγέ και μόνο με συνεργασία μπορούμε να το επιτύχουμε. Μόνο, ξαναλέω, με συνεργασία και όχι με μια ε, ε, προσέγγιση ε, ελεύθερη και ωραία, να το πω έτσι εντό εισαγωγικών. Μιλούμε για νομοθεσία. Ε, πιστεύω ότι η νομοθεσία κάποτε θα θεσπιστεί. Θέλουμε να δούμε νομοθεσία η οποία να μην είναι ξεχωριστή αναχώρα. Θέλουμε να είναι μια νομοθεσία η οποία θα προσφέρει ίσους όρους ανταγωνισμού, αλλά θα κάνει όλες και όλους μας να κατανοήσουμε τι είναι αναγκαίο για κάθε μια χώρα το γερμανικό ή το ολλανδικό παράδειγμα δείχνουν πώς μπορούν κάποια πράγματα να παράγονται τοπικά, όμως μετά να γίνει το συντονισμό σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Και για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε τέτοιου είδους συμφωνίες. Αλλά, ξαναλέω, συντονισμένες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Διακόπτη η Λίντα Μακάβαν. Το μήνυμά σας λοιπόν είναι ότι η επιχείρησή σας αναμένει νομοθεσία. Και αυτό είναι καλύτερο και για εσάς, γιατί έχετε τότε στην πραγματικότητα αυτή ε, ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Δεν ε, μπορούν δηλαδή να σας ε, ανταγωνιστούν με, κατεβάζοντας τα, τα, πρότυπα κάποιες, κάποιοι άλλοι ανταγωνιστές σας. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το επίπεδο ισότιμου ανταγωνισμού. Θα επανέλθω στη Μαριέτα, διότι νομίζω ότι οι περισσότερες, ώρες, περισσότερες ερωτήσεις ήταν για σας. Ναι, θυμούμε, ναι, μεγάλη πρωτοβουλία από τη ε, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ και μετά αποδυναμώθηκε κτλ. Τέλο πάντων δεν ήταν αυτό που αναμέναμε. Έχει γίνει λοιπόν πρόοδος. Και μετά θα αναμένω από εσά και συστάσεις για το τι μπορούν να κάνουν οι συνάδελφοί μας και η επόμενη Επιτροπή. Μαριέτα. Ευχαριστώ. Ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή και ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ συνεργασίες για την ανάπτυξη προσπαθεί να εφαρμόσει αυτά που έχουμε στο έγγραφο εργασίας του προσωπικού ιδιαίτερα για να εφαρμοστούν οι οδηγίες του ΟΣΑ και για να περάσουμε από το εθελούσιο το δεσμευτικό και υποχρεωτικό και για να γίνει σωστά αυτή η μετάβαση. Τώρα για την ερώτηση για το σύμφωνο στο Μπαγκλαντές. όπου συμμετέχει η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Αμέσως μετά το ατύχημα στη Ράνα Πλάζα, ε, το 2016 εντάχθηκε και ο Καναδάς, έχουμε τακτικές συναντήσεις, η επόμενη θα γίνει τον Ιούνιο, όπου θα γίνει μια αξιολόγηση για το πώς εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και με βάση τις συμβάσεις του ILO η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. <clears throat> Μπορεί πολλοί να πούν ότι ακόμη απέχουμε πολύ από την πλήρη εφαρμογή. Υπάρχουν κάποιες επιτυχίες στο δεύτερο πυλώνα όμως. <clears throat> Ε, λοιπόν, τον Ιούνιο θα έχουμε αυτή τη συνάντηση. Θα έχουμε και ένα workshop για τις πρακτικές ε, αγορών και θα θέσουμε τα ερωτήματα. <clears throat> Με την άδεια σας κύριε Πρόεδρε να επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας τον Ιούνιο. Αν το δέχεστε. Και θα αποβάλουμε έκθεση μαζί με τον ILO <clears throat> και τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά για όλους τους πυλώνες του συμφώνου αυτού. Συζητάμε φυσικά καθημερινά με τους συναδέλφου ε, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι ψηλά και στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε τακτικά με τον Μπαγκλαντέ. Αλλά όπως ξέρετε έχουμε και μια πολύ έντονη κρίση προσφύγων στο Μπαγκλαντές που αντιμετωπίζει τον Μπαγκλαντές Και υπάρχουν και άλλα θέματα που θα τονίσει η κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ στη διάρκεια αυτού του διαλόγου. Αλλά η Κομισιόν παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό και ελπίζουμε να επανέλθουμε τον Ιούνιο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα για τις κατευθυντήριες αρχές των ΟΕΕ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε όλα τα μέλη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τηρούν αυτές τις ε, κατευθυντήριες οδηγίες κατά γράμμα και να τηρούν πλήρως και να εφαρμόζουν αυστηρά αυτές τις αρχές. Αυτό θα διευκρίνιζε πολύ καλά την κατάσταση για την ε, εφαρμογή των υποχρεώσεων των ε, συμβαλωμένων και ιδιαίτερα για τη δεύτερη φάση εφαρμογής. Τώρα, οι υποχρεωτικές προδιαγραφές. Βεβαίως, Εργαζόμαστε σκληρά για να υπάρξει αυτή η συνάντηση και με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Νομίζω πως είναι θέμα υποχρεώσεων των ΜΕΝ και των ΔΕ και θα γίνει πολύ σύντομα αυτή η συνάντηση. Θα μεταφέρω ήδη σήμερα στο γραφείο του πρώτου αντιπροέδρου το μήνυμά σας. Σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε αυτή τη βδομάδα για το πότε θα διοργανωθεί αυτή η συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Θέλουμε να υπάρχει ισοτιμία για τις εταιρείε αλλά και για τις χώρες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ε, αυστηρές προδιαγραφές για το Μαγκλαντές και μετά οι κακές πρακτικές απλώς να μετακομίσουν σε άλλες χώρες. Ένα λεπτό παρακαλώ η επόμενη. Τελικό σχόλιο. Ένα λεπτό. Μα από πού να αρχίσω λέει ο κ. Λασάλα. Οι αδυναμίες της συμφωνίας του Μαγκλαντές καλύπτει μόνο 203 εταιρείε και όχι πολλές άλλες. Ιδιαίτερα αυτές οι οποίες στέλνουν προϊόντα σε μη δυτικέ εταιρείε, στην Κίνα για παράδειγμα. Και φυσικά ισχύει μόνο για μια χώρα. Είναι μεν η δεύτερη εξαγωγική χώρα προς την Ένωση, αλλά η πρώτη είναι η Κίνα, η τρίτη είναι η Τουρκία. Στην Τουρκία έχουμε πολλά προβλήματα με την εργασία των προσφύγων, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Πολλά πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, για να υπάρξει αυτή η ισοτιμία την οποία επιζητούν διάφορες εταιρείε. Και επίσης πρέπει να γίνουν πολλά για να καταργήσουμε την καταναγκαστική εργασία και την μοντέρνα δουλεία στην αλυσίδα προμηθειών. Ευχαριστώ πολύ για το G20. Πέρυσι, υπό τη Γερμανική Προεδρία, το G20 ασχολήθηκε με τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Υπάρχει μια δήλωση των Υπουργών Εργασίας και της Απασχόλησης, περσινή, που πηγαίνει μακριά από πλευρά συστάσεων για την τήρηση των διεθνών προδιαγραφών για την προστασία των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους και το πώς θα πρέπει να συμμετέχουν και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων και τα διεθνή συνδικάτα και οι, αυτοί που κάνουν παραγγελίες Επίσης, έχουμε ένα νέο μέτρο που εγκρίθηκε στη Γαλλία για αυτούς που κάνουν παραγγελίες. Λέει πολλά, πώς να το συνοψίσω. Αυτοί που κάνουν τις κυριότερες παραγγελίες, τις μεγάλες έκτας παραγγελίες, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτό που το ΩΣΑ αποκαλεί η λογική επιμέλεια. Θα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο λοιπόν επιμέλειας συντεταγμένο, να αναφέρουν τους κινδύνους, να υπάρχουν διαδικασίες ε, τακτικής αξιολόγησης των θυγατρικών, των υπεργολάβων, των προμηθευτών, να υπάρχει δράση για τον περιορισμό των κινδύνων. Αυτή είναι η λογική επιμέλεια. Και πρέπει να υπάρχει και μηχανισμός ε, ε προειδοποίησης. Και υποχρέωση ε, παρακολούθησης της εφαρμογή των ε, ληφθέντων μέτρων. Εδώ λοιπόν προωθείται η διαφάνεια. Ο νόμος αυτός βέβαια αφορά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με κατόφλι 5.000 εργαζομένων στη Γαλλία ή 10.000 εργαζομένων παγκοσμίω. Ο νόμος αυτός θα εφαρμοστεί σε αυτούς που δίνουν ε, παραγγελίες αλλά μέσω αντανακλάσεων, αντανάκλασης θα ε, καλύψει και τους υπεργολάβους. Δηλαδή αυτός που κάνει παραγγελίες θα ζητήσει από τις συνεργαζόμενες εταιρείε να του αποστέλουν πληροφορίες για τα δικαιώματα, την υγεία των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι θα καλύψουμε την εργασία που έχει κάνει ο ΩΣΑ και όλη την εργασία που έχουμε κάνει εμεί στη Γαλλία για την ένδυση και όχι μόνο. Γιατί υπάρχει ένα γενικότερο οδηγό ε, στον ΩΣΑ για την λογική επιμέλεια που θα ανακοινωθεί 21-22 Ιουνίου στο Παγκόσμιο Φόρουμ της υπεύθυνη λειτουργία των Επιχειρήσεων. Όλες ε, λοιπόν οι κλαδικές ρυθμίσει του ΩΣΑ και αυτός ο γενικό ε, οδηγό, θα εφαρμόσει, θα βοηθήσει την εφαρμογή αυτού του γαλλικού νόμου. Ο νόμος είναι μεν σύντομο, έχει δύο-τρία άρθρα, αλλά όλα, όλες αυτές οι προδιαγραφές εξηγούν πώς πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Και ο οργανισμός μας ε, είναι μεταξύ των δυνατοτήτων ένδικων μέσων. Μέσω του τρίτου πυλώνα του ΟΣΑ οι εθνικές αρχές επαφής βεβαίως δεν είναι δικαιοδοτικές αρχές, αλλά έχουν δυνατότητα να ακούσουν παράπονα. Με συγχωρείτε, είπα πολλά. Λοιπόν,